So, since we have Mrs. here... Εφόσον έχουμε εδώ την κυρία ε, Γκούτελαντ, μπορούμε να συνεχίσουμε με το σημείο 23, την εξέταση τροπολογιών ε, για την έκθεση του πίνακα αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης το 2017. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σωστά. Αυτή η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας ε, ανταποκρίνεται στον πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα δικαιοσύνης του 2017 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 10 Απριλίου παρουσιάστηκε του προηγούμενου έτους. Ε, επειδή τα αποτελεσματικά συστήματα δικαιοσύνης ε, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη διατήρηση των αρχών στις οποίε βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πίνακα αποτελεσμάτων είναι ένα συγκρίσιμο εργαλείο για να μπορέσουν να επιτύχουν ανεξάρτητη, ποιοτική και αποτελεσματική δικαιοσύνη ε, σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο είναι ο στόχος βέβαια ενό συστήματος δικαιοσύνης. Ο πίνακα αποτελεσμάτων που ετησίως ε, δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξελιχθεί από την πρώτη φορά παρουσιάστηκε το 2013 και ελπίζω ότι θα οδηγηθούμε έτσι σε συστάσεις, θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης τους, προκειμένου να επιτύχουν το κράτος δικαίου και την αηφόρο ανάπτυξη. Η πρώτη μας συζήτηση επί του σχεδίου έκθεσης έγινε στις 22 Φεβρουαρίου. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών ε, ήταν η 6 Μαρτίου 99 τροπολογίες ε, έλαβα για ε, το σχέδιο εκθεσής μου. Σας ευχαριστώ πολύ, με ευγνώμων για τις τροπολογίες αυτές. Θα ήθελα να τονίσω κάποιες από τις βασικές πτυχές ε, των τροπολογιών. Η τροπολογία 22, 23 και 35 σκοπό έχουν να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογή του πίνακα αποτελεσμάτων στην ποινική δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι έχει νόημα, δεδομένου ότι οι προηγούμενοι πίνακες ε, αφορούσαν περισσότερο ε, την ε, επίλυση αστικών διαφορών. Για πρώτη φορά, λοιπόν, ασχοληθήκαμε με το θέμα της ποινική δικαιοσύνης. Είδαμε κάποια στοιχεία που αφορούσαν ε, τις κάποιες υποθέσεις ε, ε, εξεπλήματος χρήματος και βεβαίως ελπίζουμε ότι επειδή έχουμε, αποτελεσμα... έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα για το θέμα του ξεπλήματος ε, χρήματος, αλλά έχουμε κοινή ε, για την ποινική δικαιοσύνη. Ε, η τροπολογία 34, 36, 38 και 43 εξακολουθεί προσπαθούν ε, να δίνουν ε, ιδιαίτερη βαρύτητα στη μείωση του χάσμα των δεδομένων για κάποιους δείκτες, ε, γιατί κάποια κράτη-μέλη αρνήθηκαν να δώσουν τα στοιχεία αυτά. Η τροπολογία 95 τονίζει τη σημασία της διατήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων όσον αφορά την έγκαιρη και ταχύτατη απονομή δικαιοσύνης. Ε, άλλες τροπολογίες ε, αφορούν ε, την καλή κατάσταση του τομέα της πληροφορικής στο πλαίσιο της δικαιοσύνης που δίνει τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να αντιδρά πολύ γρηγορότερα. όσον αφορά επίσης τη δημοσίευση ε, της διαδικασίας των στοιχείων της δίκης ε, έχω λάβει τροπολογίες. Υποστηρίζω και την 54 που αφορά ε, τη διαμεσολάβηση, την 55, την 56 και την 59. Είναι ενδιαφέρουσες τροπολογίες οι οποίες αφορούν ε, κυρίως την ειδίκευση των δικαστών και το πόσο μπορεί να επηρεάσει αυτό την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του ε, συστήματος δικαιοσύνης. Θα ήθελα όμως να μάθω λίγο περισσότερα για αυτή την τροπολογία. Ε, η δίκευση των δικαστών έχει ζητηθεί σε πολλούς τομείς ε, εντό των κρατών μελών, όμως ίσως ο κύριος Ράντε, η τροπολογία 46 ε, και η κυρία Χάουτελα, τροπολογία 59 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας θα μπορούσαν να πούν λίγο περισσότερα σε σχέση με το θέμα αυτό της ε, εξειδίκευση των δικαστών. Άλλε τροπολογίε που είχαν σκοπό την ε, βελτίωση τη αποτελεσμότητα στη δικαιοσύνη και την επίλυση των διαφορών ε, αφορούσαν τους ε, πολίτες που ζουν κάτω από το ε, κατόφλι της φτώχειας ε, και, των ανθρώπων, ε, και τους ανθρώπους με αναπηρίες. Φυσικά συμφωνώ με τις τροπολογίες αυτές. Φυσικά θα ήταν καλό να διευρύνουμε τον πίνακα αποτελεσμάτων σε σχέση με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Πολλών, πολλές από τις τροπολογίες ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτούν την συλλογική ένδικη προστασία στο, πλαίσιο, να ληφθεί συλλογική προστασία στο πλαίσιο του πίνακα αποτελεσμάτων. Κάποια κράτη-μέλη είναι πιο φιλόδοξα στον τομέα αυτό, ενώ άλλα διαφωνούν. Και για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα δεδομένα ε, που αφορούν τη δικαιοσύνη και την πρόσβαση των καταναλωτών σε αυτή, ε, είναι κάτι το οποίο μακροπρόθεσμα είναι μια προϋπόθεση ε, για να υπάρχει ένα περιβάλλον που θα είναι φιλικός καταναλωτές και στους πολίτες. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια σαφή θέση σε σχέση με την ε, ύπαρξη νέων κανόνων συλλογικής ένδικης προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις, ε, 20 ε, Μαρτίου θα κάνουμε, ε, στις 29 ε, Μαρτίου συγγνώμη, θα, υπάρχουμε, θα υπάρχει μία ακόμη ε, ε, ε, ανταλλαγή απόψεων. Ελπίζω να υπάρξει μία ακόμη να υπάρξει μια ακόμη καλή συζήτηση και να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό για τις τροπολογίες αυτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ράντεφ θα πάρει πρώτος το λόγο και μετά η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ λεπτομερή ενημέρωση σε σχέση με τις ε, τροπολογίες ε, που κατατέθηκαν για την έκθεσή της. Προηγούμενες ε, συζητήσεις μας είχαν αναφερθεί και πάλι σε πολύ συγκεκριμένα θέματα επί των οποίων κατέθεσα και τροπολογίες. Ένα αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συγγνώμη, ένα αίτημα τη επιτροπή μας να ληφθεί υπόψη στον πίνακα αποτελεσμάτων η συλλογική ένδικη προστασία, όπως επίση και η ε, καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ε, πιστεύω ότι το να συμπεριληφθεί αυτή η διαδικασία θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες της Ευρώπης να έχουν μια καλύτερη προσφυγή στη δικαιοσύνη. Όσον αφορά την εισαγωγή νέων δικτών σε σχέση με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για ε, τους ΛΟΑΤ. Θα ήθελα μία ακόμη φορά να αναφερθώ ε, στην τροπολογία ε, στην οποία είχα αναφερθεί και την προηγούμενη φορά θεωρώ ότι είναι μία διάκριση κατά των υπολείπων κοινοτήτων. Δεν είναι δυνατόν να αναφέρουμε μόνο αυτή την ομάδα ανθρώπων πρέπει να είμαστε κατά της διάκρισης κάθε φύσεως, όχι μόνο ε, κατά αυτής της ομάδας ανθρώπων των ΛΟΑΤ. Ευχαριστώ. Ε, όσον αφορά την εξειδίκευση των δικαστών, εγώ συμφωνώ με αυτή την ιδέα. Πιστεύω ότι ε, πρέπει στο πλαίσιο αυτό τα κράτη-μέλη να δώσουν περισσότερες δυνατότητες ε, στους δικαστές για να μπορούν να εξειδικεύονται και σε άλλα κρατημέλη και να υπάρχει και ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης, πρέπει η δικαιοσύνη να είναι προσβάσιμη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για να είναι αποτελεσματική. Πρέπει οι αποφάσεις να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο ε, για όλα ε, τα δικαιοδοτικά όργανα ε, και ε, για τις επιχειρηματικές υποθέσεις και για τους καταναλωτές ε, και πιστεύω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση της δικαιοσύνης σε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χάουτελα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη με τη δουλειά που έχει γίνει με την κυρία Γκούτελαν θα ήθελα να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις που μου έθεσε. Οι τροπολογίες μου μαζί με τον κύριο Άντερσον 55 ε, και 59 έχουν να κάνουν με το ίδιο ζήτημα που είναι ο περίπλοκος χαρακτήρας των κοινωνιών μας και την πίεση και την ανάγκη ε, ειδικών γνώσεων που πρέπει να έχουν ε, οι δικαστές σε, αυτά, αυτό τον ραγδαία εξελιζόμενο κόσμο. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο πίνακα αποτελεσμάτων θα λαμβάνει υπόψη κάποιου δείκτε για την εξειδίκευση των δικαστηρίων με αυτό το σκοπό να υπάρχει μια πιο εξειδικευμένη γνώση ε, και να, ε, να υπάρχει καλύτερη κατανόηση των τεχνολογιών. Οι 55 και οι 59 λοιπόν ε, τροπολογίες έχουν αυτόν τον κοινό σκοπό. Χαίρομαι επίσης πολύ που η Γιούτε Γκούτελαντ είπε επίσης ότι είναι υπέρ της ενίσχυσης της ηλεκτρονικής πρόσβασης στις αποφάσεις των δικαστηρίων ώστε να συμπεριληφθεί η νομική προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Πρέπει να πω ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια φορά είχα πάει μια αποστολή στην ακτή ε, του Ελεφαντοστού και εκεί είχα ακούσει ότι πραγματικά θεωρούν ότι μια πολύ ε, ε, ευπρόσδεκτη λαϊκή θα ήταν να υπάρχει νομολογία διαθέσιμη στο διαδίκτυο ώστε να μπορούν και τα δικαστήρια ε, να ενημερώνουν καλύτερα τους πολίτες και οι πολίτες από μόνοι τους να ενημερώνονται. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σβιεύκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Χαίρομαι πολύ που συζητούμε τα αποτελέσματα αυτά σε αιτήσια βάση. Νομίζω ότι δείχνουν το κατά πόσο έχει υπάρξει βελτίωση, τι εξελίξεις υπάρχουν. Βέβαια, καλό θα ήταν να προσθεθούν κάποιες παράμετρα. και την κυρία Χάουταλα και συνειδητοποίησα ότι ενδεχομένως, δεν ξέρω τώρα, θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε έρευνα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στις ίδιες τις ε, δίκες. Δηλαδή, χρησιμοποιούν τα δικαστήρια στις δίκες, τις νέες διαδικασίες, τις νέες τεχνολογίες μάλλον. Δεν μιλώ μόνο για τη δημοσίευση της αλλά και στη διάρκεια της διαδικασίας. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν να, να υπάρξει ακρόαση των μαρτύρων εξ αποστάσεως. Επίσης, θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει όλο και στενότερη συνεργασία με τα κράτη-μέλη, με τους προσώπους του δικαστικού κλάδου. Κύριος. Με στόχο κάθε χρόνο να περιορίζεται το χάσμα, το, η έλλειψη ε, σε δεδομένα, στην πληροφόρηση. ώστε και εμείς ως πολιτικοί αλλά και οι πολίτες μας, να οι συμπολίτες μας να μπορούν πιο εύκολα να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να χρησιμοποιούν αυτό το δικαίωμα. Θα πρέπει να μειωθεί αυτό το κενό πληροφόρηση μαζί με την κυρία Μωρέν Σαφτιέ Κατέθεσα μια τροπολογία που ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ερευνά αυτά τα ζητήματα, ιδίως ό,τι αφορά τις αρπαγές παιδιών. Είναι ένα θέμα που απασχολεί την κυρία Μωρέ Σαρτιέ. Νομίζω ότι αν μιλούμε για την προσθήκη κατηγορία στο scoreboard, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε νέες κοινωνικές ομάδες. Δεν είναι καλό να εστιάζουμε μόνο σε μια κοινωνική ομάδα, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα είναι επιζήμιο προς το scoreboard. Πρέπει να σπάσουμε τους φραγμούς ε, και να καταρρύψουμε τα εμπόδια για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Θα ήθελα λοιπόν παράγραφος 12, που είναι πάρα πολύ περιοριστική και παραπλανητική ίσως τη διατύπωσή της, να αντικατασταθεί από μια άλλη διατύπωση για να έχουμε μια ευρύτερη προσέγγιση. Όπως είπε και η κυρία Γιτελάντ, Υπάρχουν 96 τροπολογίε τις έχω μελετήσει και με τις περισσότερες συμφωνώ. Νομίζω ότι συνάδουν το πνεύμα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και τη εισηγητριάς μα. Όμως υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες τι οποίε δεν θα μπορεί να στηρίξει η δική μου πολιτική ομάδα. Συγκεκριμένα αναφέρομαι τις τροπολογίες που ζητούν συμπερίληψη της ποινική νομοθεσίας, ε, του ποινικού δικαίου. Δεν μπορεί να παραμείνει τόσο γενικόλογη αυτή η διατύπωση. Το ποινικό δίκαιο δεν είναι εμπίπτη στις αρμοδίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα κάποιοι θα πούν αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει. Είναι σαν να περνάμε μια κόκκινη γραμμή. Εμείς μιλάμε για συγκεκριμένα ζητήματα, όπως είπε η συγκεκριτήρια παραδείγματος την ε, νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, που είναι ειδικά ζητήματα. Αλλά δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το ποινικό δίκαιο συνολικά θα πρέπει να ενταχθεί στο scoreboard αυτό. Γιατί ως κριτήρια μιλάμε, πού θα βασιστούμε, κοινωτικά κριτήρια δεν υπάρχουν. Αυτό ήταν κάτι επικίνδυνο λοιπόν. και θα δημιουργούσε προβλήματα στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το δικαστικό κλάδο και τα κρατημέλη εν γέννη. Θα συνιστούσα προσοχή λοιπόν. Ευχαριστώ κύριο Λεμπρετών. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Κεπτελούντα ε, που μας παρουσίασε αρκετά, με αρκετά πλήρη τρόπο τις τροπολίες που κατατέθηκαν για το σχέδιο αυτό έκθεση ότι αφορά το πίνακα αποτελεσμάτων 2017 για τη δικαιοσύνη, το λεγόμενο scoreboard. Λυπούμε που καμία από τις δικές μου τροπολογίες ε, μαζί με τη Μαρή Κριστίμπτον δεν αναφέρθηκαν, άρα δεν τις ε, θεώρησε άξιες λήψης υπόψη. Μια ε, γενική παρατήρηση. Κατ' εμέ αυτό ο πίνακας αποτελεσμάτων για τη δικαιοσύνη είναι ένα ενδιαφέρον εργαλείο. Είναι συγκριτικό εργαλείο με στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δικαστικών συστημάτων στα κράτη-μέλη. Μπορούμε λοιπόν να το αποδεχθούμε αυτό το εργαλείο. Παρότι εγώ είμαι υπέρ μιας Ευρώπης ε, που βασίζεται στην ε, συνεργασία και όχι στην επιβολή, αν θέλετε, κάποιων ε, μέτρων και διαδικασιών. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές ε, που λένε ότι θα πρέπει εθνικές δικαιοδοσίες να ε, χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν τις νέες τεχνολογίες επικοινωνών και πληροφοριών. Θετικό αυτό, πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, ό,τι έχει να κάνει με το να πείσουμε τις ε, κυβερνήσεις να έχουν μέτρα για την ε, κατάρτιση των δικασών και αυτά τα ε, μέτρα και αυτές τις προτάσεις είναι θετικές, όμως παρατηρώ ότι υπάρχουν αρκετά τμήματα του σχεδίου έκθεσης που είναι ευνοϊκά προς την Κομισιόν. Όσο περισσότερο προβάλλουμε την Κομισιόν, τόσο περισσότερο από τη συνεργασία περνάμε σε ένα είδος ολοκλήρωσης. Για το πρώτο ή υπέρ, για το δεύτερο όχι. Με την έρευνα, ναι, έχουμε καταθέσει σχετικά κάποιες τροπολογίες. Την 26, για παράδειγμα, που λέω ότι εδώ μιλάμε για εθνικά δικαστικά συστήματα, άρα πρέπει να παραμείνουν ε, εθνικά τροπολογία 37 για απαλληφή ε, το τμήμα που λέω ότι πρέπει να πέσει πλήρη σε συνεργασία με την Κομισιό. Είναι λίγο υπερβολική διατύπωση και έχουμε καταθέσει και την τροπολογία 60 για να απαλείψουμε το κομμάτι εκείνο που ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει ε, κατά κάποιο τρόπο εκ νέου ε, στην εθνική δικαιοσύνη. Υπάρχει επίσης ένα άλλο κομμάτι του κειμένου που δεν μου αρέσει, δεν θα σας εκπλήξει αυτό, εκεί που λέει ότι θα πρέπει να έχουμε ειδικού δείκτες για την πρόσβαση των ατόμων LGBTI και επανέρχομαι σε αυτό που ο Ράντεφ και επαναλαμβάνω την κριτική που εξέφρασε. Πρέπει βέβαια να καταπολεμηθούν όλου οι διακρίσει. Όχι όμω να αναφέρουμε μόνο ε, του LGBTI και να δίνουμε έμφαση σε αυτή την ομάδα, γιατί έτσι δίνουμε την εντύπωση ότι οι άλλε ομάδε δεν είναι εξίσου ε, σημαντικές για να ασχοληθούμε μαζί του. Και γι' αυτό έχουμε την τροπολογία 73 που ζητά ειδικού δείκτε για την πρόσβαση ε, στη δικαιοσύνη. Αυτό το κομμάτι που μιλάει για LGBT να διαγραφή συγκεκριμένα. Τώρα, οι δικαστέ πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από την πολιτική εξουσία. Αυτό είναι σαφέ και το υποστηρίζουμε. Άρα οι τροπολογίες που το υπενθυμίζουν ε, με βρίσκουν σύμφωνο, όμως δεν θα έπρεπε, πιστεύω, με πρόσχημα να επαναλάβουμε την επιτακτική αυτή δημοκρατική ανάγκη, η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθεί να επέμπερβολικά στο εθνικό δικαστικό σύστημα. Γιατί το εθνικό δικαιοδοτικό σύστημα είναι στοιχείο τη εθνική κυριαρχία των κρατών. Γι' αυτό επέβαλα την τροπολογία 99 με στόχο την απαλυφή ενό τμήματο του κειμένου που είναι κάπω αμφίσιμο, κάπω ασαφέ κατά την άποψή μου. Επίσης, πάντα στο πνεύμα ότι δεν πρέπει να δίνουμε τόσε πολλέ εξουσίε στην Κομισιόν. Ένα σύστημα συνεργασία ουσιαστικά υπάρχει γιατί υπάρχει ένα δίκτυο ε, πληροφόρηση που λειτουργεί πολύ καλά μεταξύ των διαφόρων ανώτατων δικαστηρίων των κρατών μελών. Αφού λοιπόν ήδη υπάρχει συνεργασία σε σεβασμό, ε, με σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας, ε, δεν είναι καλό λοιπόν να βάζουμε την Κομισιόν να παρεμβαίνει ε, κάπου που δεν είναι απαραίτητη η παρουσία της κατά την άποψή μου. Κάποια κράτη δεν δέχονται να δώσουν δεδομένα, να δώσουν στοιχεία και λυπούμε. Γι' αυτό όμω, ε, πώ εξηγείται αυτή η συμπεριφορά, ίσω από το φόβο ότι αυτό ο είναι αποτελεσμάτων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να περάσει από την απλή σύσταση στην ομή παρέμβαση και κατά λίγο αν εγκριθούν αρκετά εστροπολογίε που θα περιορίζουν το ρόλο της Κομισιόν και θα παραλαμβάνω ότι εδώ μιλάμε για την αντίδραση της συστάσης από τα κράτη και όλα αυτά που να γίνονται σε σεβασμό, με σεβασμό στην εθνική κυριαρχία, τότε θα καθησυχάσουμε τα κράτη-μέλη που δεν δίνουν ακόμη πληροφορίε και θα δείτε ότι όλα θα πάνε πολύ καλύτερα. Αυτό είναι το μήνυμα της δική μου και η δική μου άποψη και αυτή είναι και η γραμμή που διέπει τη τροπολογία τη δική μου και τη Μαρία Κριστίν. Ευχαριστώ κύριο Μαρίνιο Πίντου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ξεκινήσω ε, συγχαίροντας την εισηγήτρια για την εξαιρετική της δουλειά και κυρίως επειδή με πολύ ανοιχτό πνεύμα δέχτηκε τις διάφορες συνεισφορέ όλων των σχεδόν εισηγητών. Ήθελα να τονίσω την ανάγκη εξειδίκευσης για τους δικαστικούς λειτουργούς και τη δικαιοσύνη, γιατί η απόφαση ενός ειδικού δικαστή είναι απόφαση που έχει περισσότερη ποιότητα και περισσότερα στοιχεία που μπορεί να καθησυχάσουν την κοινωνία από την μια απόφαση που δεν είναι εξειδικευμένη τέλος πάντων που λαμβάνεται από έναν λειτουργό ο οποίος δεν είναι εξειδικευμένος. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε κίνητρα για την εξειδίκευση των δικαστών ώστε να υπάρχει καλύτερη απόδοση δικαιοσύνης και μεγαλύτερη ε, ενίσχυση της ιδιότητας του πολίτη και ε, ηρεμία στην κοινωνία η δημοσίευση και η διάθεση online των αποφάσεων, των που επιβάλλονται από τα δικαστήρια των διαφόρων κρατών μελών, είναι και αυτό μια καλή ιδέα για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, μία απόφαση, μία δικαστική απόφαση, πραγματικά ε, δίνει τις ε, επιπτώσεις της ε, που αποτρέπουν ή δίνουν κάποια κατεύθυνση, εφόσον είναι γνωστή. Όχι μόνο για τα δύο μέρη και τους δύο διαδίκους, ε, συμπεριλαμβάνει ιδεολογικά στοιχεία που μπορεί να είναι πολύ σημαντικά για όλη την κοινωνία. Υπό αυτήν την έννοια, καλό είναι να διατίθεται σε όλους τους πολίτες. Με τρόπο μάλιστα εύκολο και γρήγορο αλλά από την άλλη είναι και μια, ε, ένας τρόπος ε, να αναλάβει περισσότερες ευθύνες ε, και υπευθυνότητα ο ίδιος ο δικαστής. Δηλαδή ανάλογα με τις αρμοδιότητες του δικαστηρίου ή της ομάδας των δικαστών, η απόφαση πολλές φορές δεν είναι της ίδιας βαρύτητας όταν δεν γνωστοποιείται μπορεί να υπάρχει μια ε, προσέγγιση κάπως πιο αυθαίρετη και όχι ε, η έννοια της διακριτικής ευχέρειας στην ε, λήψη αποφάσεων από τους δικαστές. Εν τέλει, δύο παρατηρήσεις και να υποφεληθώ εδώ της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάγκη να μελετήσουμε περαιτέρω και να εμβαθύνουμε στις μεταρρυθμίσεις του δικαστικού συστήματος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό την έννοια ότι η ίδια η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι πραγματική ολοκλήρωση εάν βασιστούμε μόνο στις εμπορικές, οικονομικές και τραπεζικές πτυχές. Πρέπει, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, να σκεφτούμε τι είναι εγκληματική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι κάτι μπορεί να θεωρηθεί εγκληματική ενέργεια στο Βέλγιο και κάτι άλλο στην Πορτογαλία ε, και η δικαστική λειτουργία να μετακινούνται από χώρα σε χώρα, οι κατηγορούμενοι, οι ένοχοι, το ίδιο. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε αυτή την επικίνδυνη και πολύ επίκαιρη διάσταση της ε, ανάμειξης πολιτικής δραστηριότητα με τη δικαστική, την αποδόση της δικαιοσύνης. Δηλαδή και επηρεάζονται πολιτικώς τα δικαστήρια και δικαστικώς επηρεάζεται η δράση των πολιτικών. Εδώ λοιπόν εμένα με τρομάζει μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι, οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορεί να διαφεύγουν από χώρα σε χώρα γιατί από τη μια κάτι μπορεί να, να θεωρείται ε, επικίνδυνη εγκληματική ενέργεια και σε μια άλλη χώρα όχι τα ίδια κριτήρια θα πρέπει να ισχύουν ε, για να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο και για να υπάρξει πραγματική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ανομοιογένεια με καταστάσεις που ζημιώνουν ιδιαίτερα την ίδια την ιδιότητα του πολίτη. Και εδώ θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον να αξιοποιήσει τις εκθέσεις μας και την αποτίμηση που έχει γίνει, την αξιολόγηση δηλαδή, το scoreboard, για να προβλέψει περαιτέρω βήματα για πραγματική ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο επίπεδο της δικαιοσύνης. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ε, does the commission wish to take... Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο. Mrs. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Να θυμίσω ότι το, ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Βαθμολογίας και Αποτελεσμάτων είναι απλώς ένα ενημερωτικό εργαλείο. Θέλει να δώσει μια επισκόπηση για τη λειτουργία των δικαστικών συστημάτων στα κάτι μελη Δεν προτείνει κάποιο ε, σύστημα δικαιοσύνης περισσότερο από κάποιο άλλο και αντιμετωπίζει ισότιμα όλα τα κράτη-μέλη στα δικαστικά του συστήματα. Το καθένα σύστημα έχει να κάνει και με την ιστορική παράδοση της κάθε χώρας και η ποιότητα καθώς και η αποτελεσματικότητα είναι η ουσιαστική παράμετρη για να κρίνουμε το αν είναι αποδοτικό ένα σύστημα δικαιοσύνη. Ε, υπό κάθε έννοια λοιπόν δεν θέλει να παρέμβει στα εθνικά δικαστικά συστήματα ο πίνακα αποτελεσμάτων. Μια επισκόπηση είναι του τι συμβαίνει. Βεβαίω, ο πίνακας αποτελεσμάτων είναι ένα ενεξελίξη εργαλείο, το οποίο το συλλάβαμε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και γι' αυτό ω τώρα ασχολείται με, με υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί ή όχι στα θέματα του εμπορικού, αστικού και διοικητικού δικαίου. Αυτό ε, το εργαλείο, όπως είπα, εξελίσσεται ακόμη και η δυνατότητα να παρουσιάσουμε δεδομένα για το πώς λειτουργούν τα συστήματα δικαιοσύνης όταν μιλάμε για περιπτώσεις διαφθοράς ή οικονομικού εγκλήματος, είναι κάτι που μας έχει απασχολήσει. Βεβαίως, όλα αυτά εξαρτώνται και από το κατά πόσο είναι διαθέσιμα τα δεδομένα στα κράτη-μέλη. Ε, κάθε μια τροπολογία που καλεί τα κράτη-μέλη να είναι πιο συνεργάσιμα για να καλυφθούν τα κενά που έχουμε στα στοιχεία είναι κάτι που το καλωσορίζουμε θερμά. Επίσης, κατά τα άλλα, οι περισσότερες τροπολογίες νομίζω ότι είναι επικοδομητικές και βελτιώνουν σίγουρα τον πίνακα αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να ε, βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων τους. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κυρία Χάουταλα. Πρόεδρε, θέλω και εγώ να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να θέσω ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την βελτίωση αυτού του τόσο σημαντικού εργαλείου. Η ερώτησή μου και δεδομένων των όσων συζητήσαμε ε, είναι περισσότερο για τις τροπολογίες, δηλαδή αυτές που αφορούν την ανάγκη να ενθαρρύνουμε και να παροτρύνουμε τους δικαστές εξειδίκευση. ή το κατά πόσο αντιλαμβάνονται οι δικαστές τι τεχνολογικέ εξελίξει, αν θα υπάρξει σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτό δεν πρέπει κάπως να ενσηματωθεί στον πίνακα αποτελεσμάτων της δικαιοσύνης. Και όπως είδατε, εδώ είναι κάπως επίμαχο θέμα για τις πολιτικές ομάδες. αν πρέπει να δώσουμε πρόσβαση ας πούμε, στη δικαιοσύνη μεγαλύτερη σε κάποιες πιο ευάλωτες ομάδες, ε, ξέρω εγώ τους Λαο ε, είναι κάτι που πρέπει να ε, συμπεριληφθεί στον πίνακα αποτελεσμάτων και δεν έχει να κάνει γενικότερα με την εφαρμογή της νομοθεσίας κατά της διακριτικής μεταχείρισης. Είναι ο πίνακας αποτελεσμάτων το κατάλληλο σημείο για να γίνει μια τέτοια ένα τέτοιο παραλληλισμό ή πρέπει να μείνει απ' έξω. Γιατί είναι ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικέ αλλαγέ. Αυτό είπαμε μόλι. Κυρία Γκούτελαντ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους ε, για τη συμμετοχή τους ε, στην επεξεργασία των τροπολογιών και για όλες τις συζητήσεις που είχαμε σε αυτό το κοινό μας ταξίδι. Ε, νομίζω ότι υπάρχει αρκετό έδαφος για να προκύψει μια άποψη συνενετική. Έχουμε και άλλες συνεδρίες σκιωδών, αλλά νομίζω ότι για τα βασικά στοιχεία της έκθεσης υπάρχει γενικώ συμφωνία. Ίσως κάποιες ε, διαφωνίες να υπάρχουν και το τι συμβαίνει με τις ευάλωτες ομάδες ή την, ε, τις συλλογικέ αποζημιώσεις και ίσως πρέπει να εμπαθύνουμε και σε κάποια άλλα σημεία, κάποιες λεπτομέρειες με τεχνικό χαρακτήρα. Ίσως έτσι δούμε το πεδίο και το εύρος του πίνακα αποτελεσμάτων για να έχει και περισσότερο νόημα, αλλά χωρίς να θέλουμε να ξεπεράσουμε και το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας ή το πεδίο που θα πρέπει να καλύπτει το, ο πίνακας αποτελεσμάτων. Απαντώντας εν μέρη, να πω ότι κάποιοι συνάδελφοι έκαναν λόγο για το πρόβλημα της στόχευσης της ομάδας των ΛΟΑΔΑ εγώ θα έλεγα ότι είναι καλύτερα να μιλήσουμε για περισσότερες ευάλωτες ομάδες και η τριοπολογία 80 αυτό κάνει. Ευχαριστώ λοιπόν τον συντάκτη ή συντάκτρια. Είναι μια τροπολογία που δείχνει ότι θέλουμε να κάνουμε περισσότερα για τις ευάλωτες ομάδες αλλά μπορεί να έχει να κάνει με το φύλλο, με τις αναπηρίες, με το σεξουαλικό προσανατολισμό, το αν ανήκει κάποιο σε βαλατη ομάδα ή όχι. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι μια καλή συμβαστική λύση και σε ό,τι αφορά, αφορά τις συλλογικές αποζημιώσεις, τις συλλογικέ προσφυγές, νομίζω ότι η βελτιωμένη πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη είναι σημαντικό και κάποιες φορές ε, έχει να κάνει και με την επιβολή του νόμου ε, σε συγκεκριμένους ε, το αστικό ή εμπορικό δίκαιο, οι συλλογικέ προσφυγές είναι σημαντικές για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο, στα δικαστήρια και να υπάρχει και επιτυχής επίλυση διαφορών. Καλό θα ήταν λοιπόν στα δικαστήρια των κρατών μελών να προβλέπονται τέτοιε δυνατότητε για συλλογικέ προσφυγές και σχετικέ δίκε. Ελπίζω να προχωρήσουμε λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση μαζί όλοι. Και μετά να ευχαριστήσω την κυρία Χάουταλα για τη διευκρίνηση που έκανε. και τις προθέσεις μας για την εξειδίκευση των δικαστών. Είναι ενδιαφέρον αυτό, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κινηθούμε μαζί, νομίζω, για να συμφωνήσουμε στο κείμενο. Νομίζω ότι η Επιτροπή απήντησε εν μέρη στην ερώτηση του κυρίου Σιδιεύκα. Και είναι ενδιαφέρον, πιστεύω, να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε το πεδίο του πίνακα αποτελεσμάτων. Θα ήθελα αυτό να γίνει βέβαια με τον κατάλληλο τρόπο, γι' αυτό θα συνεχίσω να συζητώ μαζί σα με του υπόλοιπου σκιώδει εισηγητέ και τα μέλη τη Επιτροπή Γιούρη, για να γίνει αυτό με τον καταλληλότερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ και την Επιτροπή. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα ήθελα να απαντήσω για το θέμα της εξειδίκευσης των δικαστηρίων. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της εξειδίκευσης των δικαστών, που είναι κάτι διαφορετικό από την εξειδίκευση των δικαστηρίων. Ε, αν γίνει εξειδίκευση των δικαστηρίων, υπάρχει ο κίνδυνος στα δικαστήρια να είναι πολύ ικανά για την εκδίκαση υποθέσεων ανταγωνισμού. Ε, για παράδειγμα, αν μιλάμε όμως για την εξειδίκευση των δικαστών, σημαίνει ότι δίνουμε τη δυνατότητα ε, εξειδίκευση των δικαστών σε συγκεκριμένους τομείς, αυτό μπορεί να οδηγήσει κατά τη γνώμη μου σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, γιατί δεν αφορά ολόκληρο το δικαστήριο και νομίζω ότι έτσι θα εκδικάζονται ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά οι υποθέσεις. Ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Πάμε τώρα στο 24 θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2004 ε, 35. Να περάσουμε ευθύ αμέσω στο θέμα αυτό, να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Χοακίμ Ντεουγένιο, που είναι αναπληρωτής τμήματάρχης για την συμμόρφωση και την καλύτερη ε, νομοθεσία που ε, είναι μία συνέχεια στην έκθεση της κυρίας Φεράρα. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε. Ε, χαίρομαι πολύ που θα συζητήσω μαζί σας ε, τη συνέχεια του θέματος αυτού. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας έχει ήδη ευχαριστήσει για τη δουλειά σας στο πλαίσιο αυτό, που ήταν πάρα πολύ επικοδομητική και πάρα πολύ χρήσιμη. Δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή ε, συμμερίζονται έναν κοινό στόχο, δηλαδή ότι έχουμε και συμφέρον ε, και στόχο να εφαρμόζεται σωστά αυτή η οδηγία, γιατί δημιουργεί ωφέλη, ε, πρέπει να δημιουργεί ωφέλη και ε, θετικό αντίκτυπο επιτόπου, ώστε η περιβαλλοντική καταστροφή είτε να αμβλύνεται είτε να προλαμβάνεται. Και ακόμη πιο σημαντικό, ότι η, χρήστη, η, αρχή ο, χρήστη, ο πληρώνει να τίθεται πραγματικά σε εφαρμογή. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν ζητήματα εφαρμογής, υπάρχουν κενά εφαρμογή και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει ήδη από το 2016 μια έκθεση αξιολόγησης και ήταν η βάση ε, για το ψήφισμά σα. Σχόλια και παρατηρήσεις ήταν ευπρόσδεκτα τα συζητήσαμε ε, και με τα κράτη-μέλη και από ό,τι κατάλαβα έχετε ήδη λάβει τις γραπτές μας απαντήσεις ε, για το ψήφισμα, ως προς το ψήφισμά σας που εξηγούν πολύ διεξοδικά τους, τα στοιχεία της δράσης που αναλαμβάνουμε, την πρόοδο που έχουμε σημειώσει και υπήρχαν και απαντήσεις σε συγκεκριμένα σημεία που είχατε καλύψει με το ψήφισμά σας. Δεν θα μπω λοιπόν σε, αυτό, σε αυτή την επτομερή διεξοδική αναφορά όλων των σημείων του κειμένου, αλλά ευχαρίστω αν έχετε ερωτήσεις να ε, απαντήσω σε ερωτήσεις που ενδεχομένως να έχετε. Σύντομα όμως θα ήθελα να σας πω ότι ο στόχος μας ευθύς εξ αρχής ήταν ε, να δούμε τα πορίσματα της ε, αξιολόγησης ε, και να τα αντιμετωπίσουμε με ένα με ένα πρόγραμμα κοινή κατανόηση σε βάση στοιχείων ε, της εφαρμογής, της ε, οδηγίας, συγγνώμη. Ε, υπάρχει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα εργασίας το οποίο το αναπτύξαμε για μια πολυετή περίοδο από το 2016. Ε, ξεκίνησε και είμαστε στο δεύτερο χρόνο εφαρμογής του. Νομίζω ότι πολλά από τα ζητήματα που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλύπτονται από το πρόγραμμα αυτό. Με πολύ χαρά λοιπόν να σας αναφέρω ότι υπήρξαν ήδη κάποια πρώτα αποτελέσματα από το πρώτο έτος ε, λειτουργίας και βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να βελτιώνεται η συλλογή δεδομένων. Ε, έχουμε μια καλύτερη κατανόηση των ε, όρων ε, που υπάρχουν στην οδηγία, όπως για παράδειγμα το κατόφλι σημασίας, significance threshold, γιατί είναι ε, κάτι το οποίο ε, ήταν αντικείμενο μεγάλης ανησυχίας. Ένα από τα θέματα που εξακολουθούν να υφίστανται είναι ότι απέχουμε ακόμη πολύ από μία ε, καλή κατανόηση της εφαρμογής της Οδηγία αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε σχέση με την ε, εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων. Έχουμε αρχίσει λοιπόν να συλλέγουμε δεδομένα και από πηγέ άλλε εκτό των κρατών μελών. Έχουμε έρθει σε επαφή με μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, με επιχειρηματίε, να δούμε τι άλλα δεδομένα μπορούμε να βρούμε για να έχουμε μια καλύτερη αίσθηση του τι συμβαίνει. Και έτσι ίσως να μπορέσουμε καλύτερα να, να καταλάβουμε πώς αντιμετωπίζει ε, κάποια προβλήματα περιβαλλοντικά το κάθε κράτος μέλος υπό τη συγκεκριμένη οδηγία που συζητούμε ή υπό την εθνική νομοθεσία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να καταγράψουμε αυτήν την συλλογή πληροφοριών και να αναπτύξουμε ε, δελτία αναχώρα μέχρι το τέλος του έτους. Και μετά θα τα μοιραστούμε και μαζί σας βέβαια. Δεν πιστεύουμε ότι έτσι θα καλύψουμε τα πάντα, όλα τα κενά, αλλά πιστεύουμε ότι είναι ένα καλό βήμα για μια καλύτερη, προς μια καλύτερη εικόνα. Δεύτερο στοιχείο, θέλουμε αυτή τη συλλογή στοιχείων να τη χρησιμοποιήσουμε ε, όχι μόνο για καλύτερη κατανόηση, αλλά για να πούμε σε διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με τα κράτη-μέλη σε σχέση με ε, την αιτήσια... Ε, αξιολόγηση εφαρμογής. Ε, πρώτη τέτοια αξιολόγηση έγινε το 2017. Υπήρχαν αναχώρα συστάσει σε σχέση με την οδηγία περιβαλλοντικής ευθύνη και έχουν να κάνουν από τη μία με την ύπαρξη ενός μητρώου ε, περιπτώσεων και από την άλλη να δούμε κάποιε κάποιες που υπάρχουν στο σύστημα χρηματοδότηση. Βέβαια, έχει περάσει ένα χρόνο, γίνεται ήδη ένα απολογισμό, του τι έχουν κάνει τα και ο στόχος μας είναι να γίνει ένας δεύτερος γύρος εθνικών αξιολογήσεων ε, υπό την αξιολόγηση, την αξιολόγηση εφαρμογής ε, ε, και για να καλύψουμε την νομοθεσία περιβαλλοντικής ευθύνης, αλλά και να υποβάλουμε και νέες συστάσεις για το μέλλον. Κάτι ακόμη που θα ήθελα να πω είναι ξέρουμε ότι η βάση αυτή όλων αυτών των στοιχείων είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν αυτά τα στοιχεία ε, γιατί όπως γνωρίζετε η οδηγία περιβαλλοντικής ευθύνης ε, δεν ε, περιέχει διάταξη που να υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να το κάνουν αυτό. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα εξετάζει κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μια τροποποίηση ε, ως συνέχεια της δουλειάς μας και για τη βελτίωση της, περιβαλλοντικής, της ε, υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων να, να υπάρξουν κάποιες συστάσεις σε σχέση με τη συλλογή των στοιχείων αυτών για την ε, οδηγία περιβαλλοντικής ευθύνης από τα κράτη-μέλη. ελπίζουμε να υπάρξει μια νομοθετική πρόταση το Μάιο ή τον Ιούνιο από πλευράς μας. Αυτή είναι η, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμά μας, αλλά δεν έχουμε ακόμη αποφασίσει για το πεδίο εφαρμογής και το, ε, το πώς και αν θα καλύπτεται η συγκεκριμένη οδηγία. Γιατί υπάρχουν ε, κάποια προβλήματα, κάποιες προκλήσεις νομικής ε, φύσεως και πρακτικής φύσεως που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Στο ψήφισμα αναφερθήκατε επίσης στην ανάγκη περισσότερων επιθεωρήσεων Εν μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρότεινε ένα σχέδιο δράσης ε, για τα περιβαλλοντικά θέματα και κατά τη γνώμη μας καλύπτει τα, τις περισσότερες ανησυχίες και τα ζητήματα που είχε θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα και αναφέρομαι κυρίως στην ε, παράγραφο 35 του ψηφισματός σας. Και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, Υπάρχει πλέον και ένα σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στα περιβαλλοντικά ε, θέματα από τον Απρίλιο του 2017. Και στην παράγραφο 48 του ψηφίσματός σας ε, τονίζεται και πάλι την ανάγκη ε, περισσότερων μέσων και περισσότερης δουλειάς ως προς το σημείο αυτό. Και αυτό κάνουμε αξιολογούμε την κατάσταση στα κράτη-μέλη και θα το κάνουμε μέσω αυτής της ετήσιας αξιολόγησης ε, και θα δούμε κατά πόσο θα λάβουμε άλλα μέτρα ε, για το συγκεκριμένο θέμα. Ε, αν... Εγώ ήθελα αυτά σε πρώτη φάση να σας πω ως πρώτη απάντηση να ολοκληρώσω ευχαριστώντας σας για το ενδιαφέρον σας και για την συνεισφορά σας ε, στην εφαρμογή της οδηγίας περιβαλλοντικής ευθύνης. Με χαρά θα συνεργαστούμε μαζί σας περαιτέρω, γιατί ο κοινός μας στόχος είναι ε, βέβαια το να λειτουργεί σωστά αυτή η οδηγία υπέρ των πολιτών μας. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως εισηγήτρια της ε, έκθεσης του Κοινοβουλίου για την ε, περιβαλλοντική ευθύνη και την πρόληψη των ζημιών από λόγους περιβαλλοντικούς θα πρέπει να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την εξακολούθηση στο θέμα που έδωσε η οποία όμως δυστυχώς δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες του Κοινοβουλίου. Πέραν από κάποιες διευκρινήσεις που μας δώσατε για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επεκφύγατε των βασικών ε, ζητημάτων που θέτει η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου. Κατά πρώτον, την κατεπίγουσα ανάγκη να ξεκινήσει η αναθεώρηση της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη ε, και να φανεί ότι μπορεί να υπάρξει και κάποια πολιτική λύση στα θέματα που έθεσε το Κοινοβούλιο. Εκτιμούμε βεβαίω την προσπάθεια που καταβάλλεται για να επιβληθούν κυρώσει ε, στα κατημέλη που δεν συμμορφώνονται με τι οδηγίε, όπω και το σχεδιασμό που οδήγησε στην αναδιατύπωση και το πολιτέ πρόγραμμα 2017-2020. Επίση, εκτιμούμε το κοινό έγγραφο κατανόηση για του ορισμού και τι έννοιε τη οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη και όλα τα υπόλοιπα μέτρα που προγραμματίζονται για την ενημέρωση και την κατάρτιση. Επί της ουσίας όμως αυτά τα γνωρίζαμε. Πέραν από κάποιες συγκεκριμένες σκέψεις τις οποίες ε, ταυτιζόμαστε στις απόψεις μας, φαίνονται και στην έκθεση του Κοινοβουλίου, στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν βρήκα τίποτε που επί της ουσίας να λύνει τα προβλήματα ως προς τα περίπλοκα θέματα που θέτει και το ψήφισμα το οποίο υπήρξε στη Θα θέλαμε να τα, να τα μελετήσουμε σημείο προς σημείο τι απαντήσεις δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο, γιατί καταρχήν ζητήσαμε αναθεώρηση της οδηγίας ε, περιβαλλοντικής ευθύνης, κυρίως ε, την, ε, τον νέο ορισμό της περιβαλλοντικής ζημίας. Όμως είπαμε ότι αυτό το δούμε μετά την ολοκλήρωση του πολιετούς προγράμματος από το 2017 ως το 2020 και ότι την ερχόμενη τριετία μπορεί να έχει συγκεντρωθεί απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη για να προγραμματιστεί μια αναθεώρηση. Υπ' αυτήν την έννοια όμω εμεί ελπίζαμε ότι αναθεώρηση θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο γρήγορα. Κυρίως ε, λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια σημασία που έχει η έννοια τη περιβαλλοντική ζημίας. Διότι μπορεί Εάν ξεκινήσουμε τα 4-5 χρόνια τις σχετικέ εργασίες, να συνεχίσουμε να έχουμε ω σημείο αναφοράς έναν ορισμό ο οποίο έχει φανεί και έχει αποδειχθεί ότι ήταν ε, ελλειπής. Ω δεύτερο σημείο εκφράζουμε την ε, δυσαρέσκειά μας για το δύσκολο ορισμό τη ε, τιμή της ε, σχετικής τιμής. Το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας πει ως το 2020-2021, σε τέσσερα πάλι πέντε χρόνια δηλαδή, πότε μπορεί να τροποποιηθεί η έννοια αυτή. Το ίδιο ισχύει και για το αίτημα να δοθεί, μια πιο σαφής, να δοθεί ένας πιο σαφής ορισμός για τον γεωγραφικό ορισμό που απαιτείται από την, περιβαλλοντική, από την Οδηγία Περιβαλλοντικής Ευθύνης για το ευνοϊκό καθεστώς. Επίσης για την περιβαλλοντική ευθύνη και τις ζημιές σε πρόσωπα ή σε περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει τελείω αυτή την πιθανότητα και θεωρεί ότι είναι απερχιωμένα μοντέλα όπως ο ρηπαίνων πληρώνει που ισχύουν για την αυτοκινητοβιομηχανία είναι προτιμότερα. Δεν γίνεται πάντοτε όμως κάτι τέτοιο. Σκεφτείτε τι γίνεται με μια πυρκαγιά. Α σκεφτούμε ότι μπορεί να πιάσει πυρκαγιά ένα χώρο αποκομιδή ε, απορριμμάτων όπως έγινε στη χώρα μου την Ιταλία τους προηγούμενους μήνες. Στην περίπτωση αυτή τι θα πρέπει να φορολογηθεί, τι αποζημίωση μπορεί να δοθεί στο περιβάλλον και στους πολίτες. Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί κάποια αποζημίωση να επιλύσουν τα προβλήματα που έχουν προκληθεί και στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων. Αυτά μάλιστα έχουν κοινωνικό κόστος πολύ μεγαλύτερο από τις διάφορες αποζημιώσεις που μπορεί να πληρωθούν. Και γιατί είδους φόρους μιλάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, μιλάμε για συγκεκριμένο φόρο όπως αυτός που ανέφερα εγώ. Ε, και επαναλαμβάνω, αυτά πληρώνονται είτε στα εθνικά υγειονομικά συστήματα ή ε, πολλές φορές το τίμημα το αναλαμβάνουν οι ίδιοι πολίτες στο πετσί τους. Υπάρχει και το θέμα της αστικής ευθύνης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει διάκριση μεταξύ αυτής της ευθύνης και της περιβαλλοντικής. Όμως, μιας και μιλάμε για την αστική ευθύνη, αυτό που μας λέτε δεν μας ικανοποιεί. Διότι λείπει ο ορισμός της περιβαλλοντικής ζημίας που να συμπεριλαμβάνει την ε, επιδείνωση της υγείας. Αυτό σημαίνει ότι επειδή δεν υπάρχει νομική βάση, δεν μπορούν και οι πολίτες να προστατευτούν και να, αποδει... να αποδειχθεί ε, ο συσχετισμός ε, της επιδείνωσης της υγείας τους με μια περιβαλλοντική καταστροφή. Ε, επίσης, το αίτημά μας να υπάρχει κάποια υποχρεωτική οικονομική εγγύηση, όπως να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Προστασία του Περιβάλλοντος και τις ζημιές που έχουν προκληθεί από την βιομηχανική δραστηριότητα που έχουν να κάνουν με την περιβαλλοντική ευθύνη, αυτό θα έλυνε τα προβλήματα που δημιουργούνται όταν λόγω χάρη μια εταιρεία πτωχεύει ξαϊλώνεται και δεν ξέρει κανείς ποιος έχει την ευθύνη. Δεν υπάρχει τρόπος να αποδοθεί ευθύνη. Ούτε να υπάρξει πληρωμή, ούτε αποζημίωση ε, για όποιον έχει πληγεί ε, και έχει υποστεί ζημιά από αυτό που προκλήθηκε, που προξενήθηκε. Η ρήπανση μόλις παραμένει και κανείς δεν πληρώνει. Οπότε πάλι ανατρέπεται η αρχή ο πληρώνει. Ε, τρίτο σημείο. Δεν κατανοούμε την απάντηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο αίτημά μα να δημιουργηθεί ένα μητρό των ε, επιχειρηματιών που έχουν επικίνδυνε δραστηριότητε. Κυρίω το σύστημα τη ε, οικονομική υπευθυνότητα που θα εγγύεται και την φερεγγιότητά του. Θα εγγυάται την φερεγγιότητά του. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα υποχρεωτικό μητρό αλλά εφόσον δεν το δέχεστε, ενίπτετε τα σχήρα σα, επιρρύπτοντα την ευθύνη και μετακινώντα την προς τα, μετατοπίζοντά την προ τα κάτι μέλη. Είναι κρίμα, διότι γίνεται ακόμη πιο δύσκολο να παρακολουθήσουμε συστηματικά το τι συμβαίνει και ακόμη πιο δύσκολο δυσχεραίνεται η δραστηριότητα της πρόληψης. Κάτι το οποίο κυρίως ε, στοχεύει η οδηγία της παραγωγικής ευθύνης. Επίσης, παραμελήθηκε τελείως η ε, δυνατότητα της φορολογικής ελάφρυνση ή άλλου είδους ανταμοιβή στις εταιρείε που λαμβάνουν μέτρα για την κάλυψη των υποχρεώσεων από την προβληματική τους ευθύνη. Ευθύνη. Ιδίω ο ορισμό ανεξαρτήτων αρχών ω αρχών έρευνα, ε, παρακολούθηση και επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης τη προβληματική ευθύνη. Λίγα είναι τα θετικά σημεία που μπορεί να σημειώσει κανεί. Είναι περισσότερο διαπιστώσει που τι περιέχει ψήφισμα του Κοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων η δέσμευση για αναθεώρηση τη πολιτική και τη νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για, για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα. Ε, αυτό εννοούσατε ίσως προηγουμένως Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν μας είπατε για νομοθετικές προτάσεις που θα έρθουν το Μάιο ή τον Ιούνιο και αν είναι έτσι παρακαλώ να μου το πείτε. Θα θέλαμε να δούμε νομοθετικές προτάσεις για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα ή αδικήματα. Ή εννοούσατε κάτι άλλο ίσως. Εν είδη ε, δεν μπορώ παρά να διαπιστώσω ότι με τη δουλειά μας, καρπό κοινή εργασίας, με συνεισηγητές από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, με τόσους συναδέλφους, σκιώδεις εισηγητές, ακροάσεις που οργανώσαμε, καταλήγουμε να έχουμε μια απάντηση και παρακολούθηση του θέματο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καθιστά κενό νόηματο ότι κάναμε. Είναι σαν να μας λέτε ότι είμαστε, δεν έχουμε νόημα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυστυχώς πρέπει να διαπιστώσουμε, ε, λίγο την όλη, το όλο θέμα, ότι το δικαίωμα πρωτοβουλίας της πρωτοβουλίας εδώ καθίσταται κενό νοήματος. Δηλαδή η, αρμοδι... η δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προτείνει νομοθετικές πρωτοβουλίες δεν έχει κανένα νόημα. Δεν μπορούμε να προωθήσουμε κανένα θέμα. Γίνεται λιγάκι γραφειοκρατικό αυτό που κάνουμε εδώ πέρα ως θεσμικό όργανο. Κάνουμε κάτι μεταξύ μας και τελικά δεν υπάρχει κανένας αντίκτυπος και καμία εξακολούθηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει λοιπόν να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι πολιτικές προτάσεις και οι νομοθετικές προτάσεις που προέρχονται από το Ευρωκοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γιάβορ, από την ΕΜΒΗ στο Συντάξιο Νομοδότησης, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την κυρία Φεράρα για την πλήρη αξιολόγηση της συνέχεια αυτής που δίνεται από την Κομισιόν. Συμφωνώ και με τη Λόρα και με την Κομισιόν. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ξέρετε σίγουρα τι θα πω εκ των προτέρων. Είναι σημαντικό όμως να το τονίσω και να το υπογραμμίσω δύο φορές. Τουλάχιστον τα σημαντικά. Ας ξεκινήσω από αυτά στα οποία είμαστε σύμφωνοι. Από την πρώτη στιγμή νομίζω ότι είχαμε μια πολύ στενή συνεργασία και κατά την άποψή μας δεν απήχαν οι απόψει μα τόσο πολύ σε ό,τι αφορά τα προβλήματα υλοποίηση οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη. Γι' αυτό και χαιρόμαστε με την έκθεση υλοποίηση και με τα συμπεράσματα, συμπεράσματα αυτή τη έκθεση που ε, δείχνει ότι υπάρχουν προβλήματα για την ε, εφαρμογή τη οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη στα κράτη-μέλη. Έχω κάποια σχόλια σήμερα σε σχέση ε, με τη δική σας παρέμβαση. Λέτε πάλι τα ίδια για τα προβλήματα υλοποίηση. Ε, δεν έχουμε δηλαδή εδώ να πούμε και πολλά, αφού συμφωνούμε τέλος πάντων. Άρα, ας ε, κάνω κάποιες ερωτήσεις. Είπατε ότι η αξιολόγηση περιβαλλοντικής εφαρμογής είναι ένα εργαλείο. Συμφωνώ ότι είναι ένα σημαντικό μέσο για να αξιολογηθεί η επίδοση του κάθε κράτους μέλους ό,τι αφορά την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Έχω όμως κάποιες αμφιβολίες ακόμη. E Στο πλαίσιο αυτής αξιολόγησης θα είναι δυνατόν πραγματικά να επιβάλλουμε την καλύτερη εφαρμογή της ε, νομοθεσίας, εφόσον ουσιαστικά πρόκειται κυρίως για συστάσεις της Κομισιόν προς τα κράτη-μέλη. Δεν βλέπω δηλαδή ε, να έχει κάποια ιδιαίτερη ισχύ αυτή η διαδικασία που θα μπορούσε έτσι η Κομισιόν μέσω αυτής να επιβάλλει στα κράτη-μέλη την καλύτερη εφαρμογή. Φυσικά έχουμε τις διαδικασίες επί παραβάση ως εναλλακτική, αλλά θα ήθελα να υπάρχει μια πιο συστημική προσέγγιση στο πλαίσιο αυτής της ε, αξιολόγησης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Πρέπει να συμφωνήσω με την κυρία Φεράρα ως προς το εξής. Τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρότερα σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις. Και δεν μιλάω μόνο για την πλημελή εφαρμογή της οδηγίας έγινε μια πλήρης αναφορά. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ εγώ στα σημαντικότερα σημεία. Το ένα είναι το πεδίο της οδηγίας. Το Κοινοβούλιο ξεκάθαρα ζητά από την Κομισιό να αναθεωρήσει την οδηγία της περιβαλλοντικής ευθύνης σε ό,τι αυτό το πεδίο εφαρμογή για να συμπεριληφθεί ατμοσφαιρική ρήπανση, για παράδειγμα και άλλα που δεν περιλαμβάνονται. Είχαμε επίσης κάποιες ερωτήσεις για τους ορισμούς στην οδηγία. Τώρα για την αναθεώρηση μέχρι το 23. Εντάξει, να μην πω ότι είναι απαράδεκτο, γιατί ό,τι γίνει αποδεκτό είναι τελικά, αλλά τέλος πάντων είναι πάρα πολύ λυπηρό που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί γρήγορα να προβεί στην αναθεώρηση τη οδηγία για να συμπεριλάβει κάποια στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά. Κάτι ακόμη πολύ σημαντικό είναι τα συστήματα οικονομικής ε, ευθύνης. Αν δεν είναι υποχρεωτικά αυτά τα προγράμματα, τότε η αρχή ορυπαίνων πληρώνει, μένει στα χαρτιά. Και δεν γίνεται πραγματικότητα στα κρατημέλη. Εδώ λοιπόν αυτό που ξεκάθαρα χρειάζεται είναι η αναθεώρηση της οδηγίας ώστε να υποχρεώσει σε σύναψη ασφαλήσεων ε, ε, για τα περιβαλλοντικά ζητήματα ώστε τελικά να πληρώνει ο ρηπαίνων. Πρέπει να υποχρεωτικά αυτά τα στήματα να είναι πλήρη, συνεκτικά και να δημιουργούν στην Ευρώπη τελικά ένα σύστημα όπου στα κράτη-μέλη το επίπεδο προστασίας να είναι λίγο πολύ στα ίδια επίπεδα, να είναι δηλαδή ισότιμο το πεδίο ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και για τα διάφορα κράτη-μέλη. Όχι δηλαδή εύκολα κάποιοι σε κάποια κράτη να μπορούν να ρηπαίνουν το περιβάλλον, ενώ σε άλλα να πληρώνουν πάρα πολλά. Επίσης θέλουμε να προστατεύσουμε τους ε, Ευρωπαίους πολίτες με τον ίδιο τρόπο. Στα κρατημελιάρα είναι απαράδεκτο η αρχή ορυπαίνων πληρώνει σε ορισμένα κράτη-μέλη να εφαρμόζεται και σε άλλα να μην εφαρμόζεται. Τι κάνουν οι πολίτες των χωρών αυτών. Δεν έχουν την ίδια προστασία σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική ασφάλεια. Πρέπει λοιπόν εδώ το σύστημα να είναι πολύ πιο ισότιμο και ολοκληρώνοντας σας παρακαλώ να ακούσετε την έκκληση του Κοινοβουλίου και να επιταχύνετε τη διαδικασία αναθεώρησης της οδηγίας περιλαμβάνοντας τα σημαντικά αυτά ε, σημεία περιλαμβάνοντας την έκθεση. Ευχαριστώ. Thank you as well, Mrs. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεση αυτή, συνέχεια, μετά την έκθεση πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αυξηθούν οι προσπάθειε ώστε η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη να αποδώσει όπω θα έπρεπε. Πολλά από όσα είπε ο συνάδελφο μου είναι κοινά και εγώ έχω τους ίδιους φόβους και τις ίδιες ανησυχίες. Όπως είπε και η κυρία Φεράρα, το κατόφλι σημαντικότητας είναι πολύ ψηλό για να θεωρηθεί ότι πρόκειται περί περιβαλλοντική σημεία και κάποιες φορές οι ορισμοί είναι τόσο επιστημονικοί που τρέπουν διαφορετικές ερμηνείες για την περιβαλλοντική ζημία. Και έτσι και στο θέμα της ευθύνης ε, δεν υπάρχει συνεκτικότητα. Αυτό εδώ παρεκολεί και την εφαρμογή της οδηγίας στην Ένωση με ομοιόμορφο και ικανοποιητικό τρόπο όπως αναφέρθηκε και ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία. Και μιλώ για τη ρήπανση ε, και για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Συμμερίζομαι τους φόβους που ανέφεραν οι συνάδελφοι. Ότι δηλαδή Υφίσταται βλάβες ε, ε, οι συμπολίτες μας ε, λόγω της ανεπαρκούς νομοθεσίας για την προστασία της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτά υπόψη νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υποστήκατε επιγόντως να θεωρηθεί ότι για την περιβαλλοντική ευθύνη. Εμείς από πλευράς Κοινοβουλίου θα θέλαμε επίσης ο ορισμός της περιβαλλοντικής ζημίας ε, να γίνει πιο ευρύς ε, και να συμπεριλάβει περισσότερες ε, ζημίες για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη υγεία, βλάβη στην ανθρώπινη υγεία. Είπατε ότι θα καταβάλει προσπάθειες για τον ορισμό της περιβαλλοντικής βλάβης ή ζημίας η Κομισιόν πριν την αναθεώρηση της οδηγίας και μετά την αξιολόγηση REFIT 2021-2023. Όμως, θα ήθελα να μας αναφέρετε αν έχετε κάποιες πρώτες σκέψεις. Τι δηλαδή θεωρείτε ότι θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο μελλοντικό ορισμό για την περιβαλλοντική ζημία. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι και να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας εφόσον αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι το να σώσουμε ανθρώπινες ζωές από τη λίπανση. Αυτό πρέπει να γίνει. Επίσης, Ήδη μας είπατε ότι υπάρχει στην οδηγία μια διάταξη για τους μηχανισμούς λογικής ένδειξης προστασίας άρθρα 12-13. Περιβαλλοντικές ΜΚΟ, δυνάμει εθνικής νομοθεσίας μπορούν να προσφύγουν στις εθνικές αρχές για την παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τα κράτη-μέλη όμως είναι αυτά που έχουν τον πρώτο λόγο. Και αυτό θα επηρεάσει και το πώς θα κρυθούν οι υποθέσεις ε, που έχουμε μαζική βλάβη και ζημία. Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια παραδείγματα πώς η Κομισιόν σκοπεύει να βελτιώσει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και επίσης ε, τι θα περιλαμβάνει η υπερχόμενη πρόταση για τον Πανευρωπαϊκό Μηχανισμό Συλλογικής ε, Προστασίας Συλλογικών Προσφυγών. Δηλαδή θα υπάρχει δυνατότητα συλλογικών προσφυγών για περιβαλλοντική ζημία ή στην οδηγία τα ασφαλιστικά μέτρα θα είναι πιο περιορισμένο το πεδίο εφαρμογή. Θα ήθελα να πείτε τι απόψει από αυτό. commission has received a... Περίπου 50 ερωτήσεις σας, έκανε, σας κάναμε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως μπορείτε σύντομα να μας απαντήσετε ή τουλάχιστον σε κάποιες από αυτές. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, προφανώς η διεξοδική μου απάντηση δεν ήταν επαρκώς διεξοδική. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Ε, αναφερθήκατε σε πολλά ε, σημεία, αλλά δεν ε, νομίζω ότι υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ μας. Το ένα τμήμα το ένα κομμάτι, αυτό που ανέφερε ε, η συγγήτρια, ε, θα το καλύψω μετά, αλλά ε, οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ο κύριος Γιάβορ και λοιποί, ανέφεραν κάποιες προτάσεις, σημειώνουμε τις προτάσεις αυτές, πού μπορούμε να τα πάμε καλύτερα, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη δουλειά που έχει ήδη δρομολογηθεί, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των ημών και ημών. Ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το υπάρχον μέσο αυτή τη στιγμή που θα μεταγραφεί στην εθνική νομοθεσία για να υπάρξει βελτίωση. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά όλα αυτά που αναφέρατε βεβαίως θα τα σημειώσουμε και θα δούμε πώς μπορούμε να τα ε, μεταγράψουμε στην πράξη. Στις 17 Απριλίου θα ξανασυναντηθούμε με τα κράτη-μέλη και θα ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό με τα κράτη-μέλη. Θα αναφέρω στα κράτη-μέλη όλα αυτά που άκουσα εδώ σήμερα, ώστε υπό το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο να μπορούμε να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας είναι επίσης σαφές από την άλλη ότι εμείς αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε από μόνοι μας σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι πάμε στο δεύτερο τμήμα της απάντησή μου. Εκεί υπάρχει ενδεχομένως η μεγαλύτερη διάσταση απόψεων προς την ανάλυση κατάστασης. Συζητήσατε στο ψήφισμά σας ε, ρητό την ανάγκη αναθεώρησης ε, της ε, Νομοθεσία. Ε, το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει την άποψή τη από τότε, Είχαμε πει ότι πριν από την αναθεώρηση τη οδηγία πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα ποιε θα μπορούσαν να είναι οι λύσει. Γιατί η ανάλυση που άκουσα για εσά ε, σε κάποιο βαθμό μα βρίσκει σύμφωνους βέβαια, αλλά δεν συμπεριλαμβάνει τη συνδυασμένη ανάλυση με ε, τα μέσα που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Νομίζω λοιπόν ότι το είπατε κι εσείς ε, κυρία εισηγήτρια στην αρχή ότι είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα, είναι τεράστιο, γιατί δεν έχουμε ένα μέσο το οποίο πρέπει με εναρμονισμένο τρόπο να εφαρμόζεται ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια κλασική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ισχύει η επικουρικότητα και έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο, συμπληρώνει 28 εθνικά συστήματα νομοθεσίας. Και καταλαβαίνετε ότι η έννοια της ευθύνης είναι πολύ διαφορετική στα διάφορα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει λοιπόν μία ανάλυση μόνο που να μπορεί να καλύψει τα πάντα και μία λύση που να μπορεί να τα λύσει όλα. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό που πρέπει σίγουρα να κάνουμε από κοινού είναι να καταλάβουμε καλύτερα που έγινε τα προβλήματα και πώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο η νομική παρέμβαση μπορεί να λύσει το πρόβλημα με το βέλτιστο δυνατό τρόπο και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της επικουρικότητας. Εμείς ε, ε, ο στόχος μας ε, όταν συλλέγουμε τα στοιχεία είναι να υπάρχει μια καλύτερη κατανόηση, μετά να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ε, τα στοιχεία αυτά στους υπεύθυνου λήψης αποφάσεων για να αποφασίσουν αν ο καλύτερος τρόπος να βελτιώσουμε την κατάσταση είναι μέσω της αναθεώρησης ή όχι. Εμείς λοιπόν τώρα συλλέγουμε στοιχεία για την ώρα και θα δούμε στο μέλλον πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή υπήρχε για τα συστήματα, για τα προγράμματα χρηματοοικονομικής ασφάλειας, ε, είδαμε ότι σε μερικα κρατημέλη λειτουργούν πάρα πολύ καλά και είδαμε τώρα ότι μπορούμε να, να δημιουργήσουμε και άλλα τέτοια προγράμματα σε κάποια άλλη... άλλα γιατί θα τους ήταν χρήσιμο. Νομίζω λοιπόν, και αυτό το λέω ως παράδειγμα για να σας εξηγήσω, ότι είναι ε, πολύ σημαντικό πριν κάνουμε μία αλλαγή σε νομικό επίπεδο πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η αλλαγή σε επίπεδο νομοθεσίας ε, επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Εμείς παντούς για την ώρα δεν έχουμε πρόθεση να ξεκινήσουμε αναθεώρηση της οδηγίας. Για την ώρα σημειώνουμε λοιπόν αυτή τη διάσταση απόψε, αλλά δεν σημαίνει ότι για αυτό το λόγο δεν μπορούμε να συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα θέματα που αναφέρατε. Για μένα είναι σημαντικό να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη, με ε, την κοινωνία των πολιτών, με τον κλάδο, δεν προσπαθούμε να κρυφτούμε πίσω από τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να βγούμε να ψάχνουμε τα στοιχεία που θέλουμε να συλλέξουμε χωρίς τη βοήθεια των κρατών μελών. Και ε, πρέπει να υπάρχει και ένα σύστημα που να επιτρέψει τη δημιουργία ενός μητρώου. Μπορεί να μην χρειάζεται λοιπόν μια νομική απέτηση για να δημιουργηθεί ένα μητρό. Μπορούμε να αρχίσουμε να συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα στα διάφορα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων μάλιστα υπήρξαν και ορισμένα που ε, το κάνουν ήδη. Ε, είναι δημόσια τα δεδομένα αυτά και δείχνουν πώς αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά ε, Περιβαλλοντική ευθύνη σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ να ξανασυζητήσουμε μαζί σας το θέμα αυτό και να σας αναφέρουμε οποιαδήποτε πρόοδο στη συνεργασία μας με τα κράτη-μέλη και αν έχετε ε, βεβαίως ε, οποιαδήποτε πληροφορία για κάποιες λύσεις που θα μπορούσαμε να βρούμε επί των σημείων που αναφέρετε, ευχαριστώ να τα ακούσουμε γιατί κάθε φορά που σκεφτόμαστε την αναθεώρηση τη οδηγία αυτή στο μέλλον, ε, σκεφτόμαστε ότι πρέπει να είναι ε, τέτοια αναθεώρηση ώστε σε πέντε χρόνια να μην έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα και να ε, μην μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν για την οδηγία της του περιβαλλοντικού εγκλήματος αυτό είναι βέβαια αντικείμενο ε, αναθεώρησης αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε όμως αν θα χρειαστεί αναθεώρηση της οδηγίας ακόμη. Το εξετάζουμε. Και επίσης πρέπει να δούμε και την ε, ε, ε, υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Κάνουμε λοιπόν έναν έλεγχο καταλληλότητας για να δούμε κατά πόσο η περιβαλλοντική νομοθεσία μπορούσε να υποφεληθεί από την ενίσχυση των δεδομένων που θα επιφέρουν τα τα προγράμματα αυτά συλλογής δεδομένων στα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι το κομμάτι που δεν αφορά την ε, οδηγία για το περιβαλλοντικό έγκλημα. Ο κύριος Γιάβορ επίσης είχε ε, απευθύνει κάποια ερωτήματα, αλλά εφόσον έφυγε θα τα πω διμερώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Αυτά για το σημείο 24 της ημερησίας διάταξης. Να σας ενημερώσω απλώς ότι το επόμενο, η επόμενη συνεδρίασή μας θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες ε, τη Δευτέρα 23 Απριλίου από τις 3 το απόγευμα ως 6.30 και στις 24 Απριλίου, ημέρα Τρίτη, να σας υπενθυμίσω επίσης ότι θα υπάρξει μια κοινή ε, συνεδρίαση με την Επιτροπή Συνταγματικών, ε, την ΑΦΚΟ. Ε, έχει προγραμματιστεί για αύριο, 28 Μαρτίου, από τις 11.30 στις 12.30. Στην αίθουσα ASP 3Y2. Ελπίζω ότι θα βρεθούμε εκεί και ότι θα προσέλθετε. Αν όχι, καλό Πάσχα. Εύχομαι σε όλους.